σε τρίτες χώρες. Το λόγο έχει εισηγείται για τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα παραποιημένα ε, προϊόντα είναι επιζήμιοι για τους καταναλωτές και βάλουν κατά της οικονομίας, της ποιότητας και της έρευνας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια στρατηγική για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Μια στρατηγική η οποία πραγματικά να μας δίνει μεγαλύτερη προσβασιμότητα σε κάποια ευαίσθητα προϊόντα όπως τα φάρμακα. Οι βασικές αυτές αρχές διέπουν αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας όσον αφορά τη στρατηγική για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες. Έκθεση η οποία στις 14 Απριλίου εγκρίθηκε από την Επιτροπή μου την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου και ανταποκριθήκαμε κατά αυτόν τον τρόπο στην ανακοίνωση του Ιουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ιουλίου 2014, προκειμένου να έχουμε μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική μετά την κατάρρευση της συμφωνίας Άκτα. Τα δικαιώματα διανοητική ιδιοκτησία έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία δέκα χρόνια, ακριβώ επειδή αλλάζουν πάρα πολύ οι τεχνολογίε, χρησιμοποιούνται νέε τεχνολογικέ καινοτομίε ακόμα και στι αναπτυσσόμενε χώρε. Γι' αυτό ακριβώ το το λόγο χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική στρατηγική, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις και θα πρέπει να προτείνει συγκεκριμένε ε, συνεπείς παρεμβάσεις. Το 39% της οικονομικής, συνολικής οικονομικής δραστηριότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα 26% των θέσεων απασχόλησης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούνται από υπηρεσίες οι οποίες ε, επενδύουν σε δικαιώματα διοντικής διοκτησίας ή επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δικαιώματα διοντικής διοκτησίας. Την πρόταση που παρουσιάζουμε λοιπόν σήμερα και που θα εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολουθούμε ουσιαστικά την προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί θεωρούμε ότι η προσέγγιση αυτή είναι καλά ισορροπημένη και αντανακλά διάφορε αποκλίνουσε προσεγγίσει και αποκλίνοντα συμφέροντα. Του χρήστε από τη μια, του καταναλωτέ και του δημιουργού από την άλλη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία νομοθεσία η να λειτουργεί καλά αν πραγματικά δεν εμπλέκονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορεί. Ένα λόγο παραπάνω λοιπόν προκειμένου προκειμένου να καταφέρουμε και εμείς τη δική μας στρατηγική να εμπλέξουμε όλους τους πολίτες οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς πώς λειτουργούν τα δικαιώματα διοντικής διοκτησίας και θα πρέπει να αναλάβουν μία υπεύθυνη στάση ιδίω απέναντι στα παραποιημένα προϊόντα και τα προϊόντα πειρατεία. Δεν θα πρέπει τα δικαιώματα διοντικής διοκτησία και η πειρατεία να θεωρούμε ότι αφορά μόνο τα προϊόντα πολυτελείας. Αντίθετα, αφορά πολλές φορές τα φάρμακα, τα καλλιντικά, τα ίδια τα παιχνίδια. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, εμπλακούν, να εμπλακεί όλο και περισσότερο και να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια συντονισμό σε όλε τι δράσει τι οποίε εγκρίνει. Αν περάσουμε περισσότερο στι λεπτομέρειε, σα έλεγα ότι τα βασικά στοιχεία τη έκθεσή μου είναι ότι θα πρέπει καταρχά να γίνει μία διάκριση ανάμεσα στην παραποίηση προϊόντων και την παραβίαση των διονετικών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερο συντονισμό με τι ελληνικέ αρχέ, ένα καλύτερο επικοδομητικό διάλογο προκειμένου να εμπλακούν όλοι οι αναφερόμενοι φορεί. Πρέπει από την άλλη να ενισχύσουμε το παρατηρητήριο το ευρωπαϊκό για την παραβίαση των δικαιωμάτων διοντική διοκτησία. Το παρατηρητήριο αυτό θα πρέπει να είναι εντελώ ανεξάρτητο. Θα πρέπει να έχουμε προσιτέ τιμέ όσον αφορά τα γενώσιμα φάρμακα, ιδίω για τι τρίτε αυτέ χώρε τι οποίε προωθούνται, προκειμένου να μπορούν όλοι οι πολίτε να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα αυτά. Πρέπει επίση να πούμε ότι οι γεωγραφικέ ενδείξει είναι πάρα πολύ σημαντικέ, όπω και τα υπόλοιπα δικαιώματα διοντική διοκτησία γιατί μέσω των γεωγραφικών ενδείξεων μπορούμε πραγματικά να έχουμε ένα σύστημα εχνηλασιμότητα για συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία πάνε προ καταναλωτέ και προστεύουμε περισσότερο του παραγωγού. Επίση, θέλουμε να προωθήσουμε ένα κέντρο εξυπηρέτηση, help desk, ιδίω όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων διανοητική διοκτησία στι τρίτε χώρε. Θεωρώ ότι η έκθεση αυτή αποτελεί ένα πρώτο βήμα θετικό, στο οποίο όμω θα πρέπει να, να, το οποίο θα πρέπει να επεξεργαστούμε ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Θα πρέπει να καταφέρουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά τις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες οι οποίες συνάπτουμε με τρίτες χώρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε στη διαδικασία του ΚΑΤΣΔΙ. Κύριε Σοντζουλίτσα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λαμβάνοντα υπόψη τι σημαντικές αλλαγές οι οποίες έχουν λάβει η χώρα στον τομέα της πνευματική ιδιοκτησία τα τελευταία χρόνια, πιστεύω ότι η προστασία και η εφαρμογή των ε, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησία είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να αντιμετωπίσουμε την ε, απειλή της πειρατείας ε, σε σχέση με την ευρωπαϊκή δημιουργική βιομηχανία, τις θέση απασχόλησης και την ανάπτυξη. Ξεπεράστηκαν τα προβλήματα με την άκτα η οποία αντιμετώπιζε την προστασία του ίντερνετ μαζί με την προστασία της πνευματική ιδιοκτησίας. Νομίζω ότι μια σωστή προσέγγιση είναι αυτή που αντιμετωπίζει και τα θέματα διανοητικής ε, ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν παγκόσμιοι κανόνες για το, τη διανοητική ιδιοκτωσία. Επίσης νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό πρέπει να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των γενώσιμων φαρμάκων που εξασφαλίζει και την έρευνα αλλά και την ε, πρόσβαση σε φαρμακείο. Μαριά. Κύριε Πρόεδρε, η ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίζεται όχι στη μείωση των μισθών, αλλά στην καινοτομία και στην οικονομία τη γνώση. Οι κλάδοι ένταση δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία παράγουν το 39% τη συνολική οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αξίας 4,7 επτά τρισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως και απασχολούν το 26% του συνολικού εργατικού δυναμικού δηλαδή 56 εκατομμύρια εργαζόμενους. επομένως απαιτείται ένα πλαίσιο νομικής προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας όχι μόνο στην ευρωπαϊκή ένωση αλλά και στις τρίτες χώρες. ταυτόχρονα πρέπει να ανατραπεί η κατάχρηση δικαιώματος εκ μέρους των κατόχων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και να ανατραπεί η δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων εκμετάλλευσης και αισχροκέρδειας ειδικότερα σε σχέση με τις φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες ενεργώντας κατά κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους έχουν μετατρέψει την εμπορία φαρμάκων σε μια αισχροκερδή επιχείρηση συσσόρευσης υπερκερδών σε βάρος των τρίτων χωρών οι τιμές των φαρμάκων πρέπει να είναι προσιτές στους στοχοποιημένους λαούς της ευρώπης και των τρίτων χωρών γιατί η υγεία είναι δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει καμιά αφεβολία ότι η παγκοσμιοποίηση έφερε πολλά θετικά στον πλανήτη μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος λοιπόν να μην στηρίξουμε την Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και τα ωφέλη από το παγκόσμιο εμπόριο. Όμως η παγκοσμιοποίηση δημιούργησε και πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, απομίμηση προϊόντων, πλαστά προϊόντα δηλαδή. και μάλιστα βοηθάει πολύ το ηλεκτρονικό εμπόριο για να πουλούνται τέτοια προϊόντα. Εμείς λοιπόν πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες εκείνες που θέλουν να προστατεύσουν την ε, διανοητική ιδιοκτησία. Τα παραπημένα, οι απομιμήσεις δεν οδηγούν μόνο σε ωραίες τσάντες και τέτοια προϊόντα, οδηγούν και σε πράγματα που μπορεί να βλάψουν την υγεία μας. Πλαστά φάρμακα για παράδειγμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τώρα πέντε λεπτά συζητάει το Κοινοβούλιο πριν συνοψίσει η Επίτροπος. Λοιπόν, πώ είναι δυνατόν να κάνουμε σοβαρά μια τέτοια συζήτηση. Εγώ διάβασα τι 14 σελίδε τη έκθεση αυτή και υπάρχουν δύο, δύο λέξει που δεν βρήκα πουθενά. Μικρέ επιχειρήσει. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα με τα δικαιώματα διανοτική ιδιοκτησία είναι ότι μικρέ επιχειρήσει δεν μπορούν να ε, ακολουθούν τη γραφειοκρατία και να καλύψουν τις προϋποθέσεις για να μπορούν να έχουν το εμπόριό τους και να ξέρουν τι είναι πλαστό και τι δεν είναι ιδιαίτερα μάλιστα στην ψηφιακή εποχή, πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Καπούτο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα δικαιώματα διανοτικής ιδιοκτησίας ε, έχουν μία έντονη θεσμική ιστορική πτυχή και πραγματικά συνδέονται με την ίδια την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού και διεθνούς πολιτισμού. Όντως, τα δικαιώματα διοντικής διοκτησίας είναι συνειφασμένα με την ίδια την δημιουργία, με τον ίδιο τον πολιτισμό, με τον δυτικό θα έλεγα πολιτισμό και αυτό φαίνεται πάρα πολύ έντονα σήμερα γιατί η λογοτεχνική επιστημονική ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ζητήματα αλληλένδετα τα οποία βασίζονται βασικά στα δικαιώματα διοντικής ιδιοκτησίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν οι Ευρωπαίοι πολίτες να γνωρίζουν πραγματικά την βάση των δικαιωμάτων αυτών διανοητικής ιδιοκτησίας. Βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι ιδίως όσον αφορά τον τομέα των φαρμάκων υπάρχει μία άδειλη, σκιώδης οικονομία η οποία λειτουργεί εντελώς αρνητικά και πολλές φορές οδηγεί στην παραγωγή αυτών των παραποιημένων φαρμάκων. Βλέπουμε λοιπόν το φυστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προστατεύει ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε τις τρίτες χώρες εταίρους. Ο κύριος Τσαμπάσκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η διανοητική ιδιοκτησία έχει σήμερα τη μεγαλύτερη σημασία που είχε ποτέ στο παρελθόν. Με την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο, με τη μεγαλύτερη ψηφιακή ε, πρόσβαση που έχουν οι αναγνώστες και οι καταναλωτές πολιτιστικών αγαθών είναι ιδιαίτερα έντονο αυτό. Υπάρχουν όμως σημαντικές προκλήσεις ιδίως για χώρες οι οποίες είναι θύματα παράνομου εμπορίου γιατί δεν έχουν τους μηχανισμούς να αντιμετωπίσουν τις πειρατικές μορφές ε, των πνευματικών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα συστήματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλες τις χώρες μας. Οι χώρες που δεν έχουν πρόσβαση σε μεγάλες αγορές αντιμετωπίζουν πολλά παραποιημένα αγαθά και πρέπει να προστατεύσουμε τα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας και να ακολουθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπεγκίν για ένα λεπτό. Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζουμε σε ποια πνευματική ιδιοκτησία αναφερόμαστε. Κατά την άποψή μας η έκθεση αυτή θα μπορούσε να μας βρει σύμφωνους, αλλά περιέχει κάποια στοιχεία που μας προκαλούν ανησυχία. Το ότι, είναι αναγκαίο να επιβάλλουμε στις τρίτες χώρες τα δικά μας πρότυπα, προστασία των δικαιωμάτων διοντική ιδιοκτησία εν μέρη είναι σωστό ή μπορεί να φαίνεται σωστό, αλλά αν το κάνουμε αυτό προκειμένου να επιτρέψουμε στι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει να εγκατασταθούν στι τρίτε αυτέ χώρε για να παράγουν εκεί πέρα πιο φθηνά, τότε πραγματικά δεν ωφελούμε του Ευρωπαίου πολίτε. Επίση, τα δικαιώματα του δημιουργού στο διαδίκτυο είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα καθόδε και σε καμία περίπτωση, βέβαια, εγώ δεν προωθώ την πειρατεία, αλλά σε καμία περίπτωση επίση δεν μπορώ να δεχθώ κάποιες ε, νέες περιπτώσεις upload όπως περιγράφονται στην έκθεση αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε και μία τοποθέτηση στην έκθεση αυτή όσον αφορά το ζήτημα των φαρμάκων. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα διοντικής διοκτησίας δεν απορροφούν από την οποία κρύβουν τα συμφέροντά τους οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Γιατί νομίζω ότι αν επιτρέψουμε κάτι τέτοιο θα έχουμε χάσει μια τεράστια ευκαιρία. Ευχαριστούμε. Επίτροπος Γιώργο έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγητή την κυρία Μόσκα και την Επιτροπή που δούλεψε πάνω στην έκθεση αυτή. Η έκθεση υπογραμμίζει πόσο μεγάλη σημασία έχει η προστασία και η πρόθεση των δικαιωμάτων διανοτική ιδιοκτησία για όλου μα και για τους εταίρους μας και υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να συνεχίσει αλλά να πάει ακόμα πιο πέρα με τις προσπάθειές της προς την κατεύθυνση αυτή. Συμφωνεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, χαίρεται για την ε, εκτίμηση που δείχνεται στη στρατηγική μας όσον αφορά την προστασία και την πρόθεση των δικαιωμάτων διονοτικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες και προσπαθεί να πετύχει μια ισορροπία μεταξύ διαφορετικών συμφερόντων. Είναι σίγουρο ότι η προσπάθεια αυτή για να υπάρχει καλή η ισορροπία μεταξύ συμφερόντων των ε, χρηστών και των παρόχων είναι κάτι ιδιαίτερα περίπλοκο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλες τις πλευρές και είναι και κάτι που μας απασχολεί όλους να δούμε κάθε παραβίαση δικαιωμάτων διονοτικής ιδιοκτησίας που βλέπουμε ότι πλευρασιάζει τα τελευταία χρόνια να τιμωρείται. Και χαιρόμαστε πολύ που βλέπουμε ότι όλοι θέλετε να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Πράγματι υπάρχουν πολλά σημεία που αναφέρει η έκθεση και με τα οποία συμφωνεί απόλυτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως για παράδειγμα η ανάγκη για τα εξή. Να συμμετέχουν περισσότερο οι εμπλεκόμενοι στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, οι κυρώσεις, η συνοχή μεταξύ προστασίας τέτοιων δικαιωμάτων και επιβολής άλλων πολιτικών. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να επαναλάβουμε ότι η πρόσβαση στα φάρμακα πρέπει να γίνεται σεβαστή και να συνάδει με την προστασία των διανοητικών δικαιωμάτων. Θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι δίνουμε αρκετή σημασία και στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που έχουμε στην προστασία διονυτικών δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα αυτά, εφόσον τηρούνται και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν να βελτιώσουν την προστασία και την εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών παγκοσμίω. Παροχή βοήθειας επίσης σε τρίτες χώρες που προσπαθούν να βελτιώσουν τα συστήματά τους προστασίας διονοτικών δικαιωμάτων. Είναι και αυτό σημαντικό. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις συστάσεις της έκθεσής σας όσον αφορά την μελλοντική μας στρατηγική και την εφαρμογή των δικαιωμάτων διονοτικής διοκτησίας σε τρίτες χώρες. Προσβλέπουμε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο μέλλον και όλους τους εταίρους μας στο εγχείρημα αυτό. Θέλω να σας διαβεβαιώσω επίσης ότι όλες σας τις συστάσεις που άκουσα σήμερα θα τις μεταφέρω στη Σεσίλια Μάστρομ, τη συναδερφό μου, που είναι και η Επίτροπος Αρμόδια για το φάκελο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ και όλους εσάς αξιότιμοι προβλευτές. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Θα ψηφίσουμε αύριο στις 12 το μεσημέρι.